Ε, η ενίσχυση μιας ε, δραματικής σειράς στη Μοζαμβίκη. Ε, αυτά συμβαίνουν όταν δίνουμε χρήματα σε μια χώρα όταν ας πούμε ε, πηγαίνει σε πολλά project δωρητών ε, ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέτοια πράγματα περιμένουμε. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν απαρκείς συναλλαγές για να ελεγχθούν. Δηλαδή αυτές δεν περιλαμβάνονται στο ποσοστό σφαλμάτων. Να η ιδέα και να απλή αφού δεν μπορείτε να τα ελέγξετε, μην τα δαπανάτε. Μόνο έτσι θα βελτιώσετε τον έλεγχο του προϋπολογισμού σας. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό ο συνάδελφος Deutsch έχει το λόγο. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα πολύ σημαντικό ε, θεματοφύλακα της διαχείρισης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο εκδίδει μία έκθεση για τους λογαριασμούς της Ένωσης και αυτό αυτή η έκθεση είναι και η απαρχή της διαδικασίας απαλλαγής. Είναι η ενδέκατη φορά που ε, συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία και κατά τα διαστήματα είχα άλλη αρμοδιότητα. Να πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο κάνει εξαιρετική δουλειά, έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Τώρα για τις τάσεις να πούμε ότι η τάση είναι θετική. Δεν είναι ε, αρνητική η δήλωση αξιοπιστίας. Και τα εκτιμόμενα επίπεδα σφαλμάτων ήταν 2,6% το 2018, παρόλο που έπρεπε για κάποιες πληρωμές ε, που γίναν για επενδύσεις ε, να δοθεί μεγαλύτερη διασάφηση. Κυρία Πρόεδρε, να πω κάτι ως επικεφαλής της Ουγγρικής ε, Αντιπροσωπείας ε, στο ΕΛΚ. Θα μιλήσω στις... Ε, μπορώ να μιλάω την 23η Οκτωβρίου που είναι μια εθνική επέτειος. Θυμόμαστε την Επανάσταση του 1956, θυμόμαστε τους ήρωές μας και αυτό για μας είναι σημαντικό. Παρακαλώ, αν θέλετε να πείτε κάτι, να το πείτε μέσα στο χρόνο ε, που έχετε για να μιλήσετε. Ο συνάδελφος Φόλτερς έχει το λόγο. Για να... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τους τελευταίους μήνες Αναλωθήκαμε σε συζητήσεις για μία χώρα και μία συγκεκριμένη ερώτηση. Ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ πέρα όμως 27 ακόμα κράτη-μέλη, πέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο, που πρέπει να ασχοληθούμε με τον προπολογισμό μας για τα επόμενα 7 χρόνια. Και ο προπολογισμό αυτός, οι δημοσιονομικές αυτές προοπτικές θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια πιο φίλο περιβαλλοντική Ευρώπη και θα πρέπει να μας επιτρέψουν να λύσουμε κάποια πολύ ακαθόδη προβλήματα. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018. Πολλά τα εκατομμύρια αυτά τα οποία ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί ως πληρωμές από τα κράτη-μέλη. Πολλά τα προγράμματα τα οποία περιμένουν ακόμα να ελοποιηθούν. Προγράμματα τα οποία απεγνωσμένα χρειάζονται συγκεκριμένε περιφέρειε για να απτυχθούν περαιτέρω. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν μια προσέγγιση πιο ευφύ, να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια, προκειμένου να ελοποιηθούν προγράμματα τα οποία θα επιφέρουν προ τη θέμενη αξία στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, στον τομέα των σιδηροδρόμων. Τα επόμενα λοιπόν 7 χρόνια α διασφαλίσουμε ότι θα επεξεργαστούμε προγράμματα τα οποία θα λειτουργήσουν θετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Πίπερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ τους Βρετανούς συναδέλφου καταρχά. Με αυτές τις επιθέσεις νομίζω ότι τελικά θα διαλύσουν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ το Ελεκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εργασία Ελέγχω του προβλησμού. Είπατε 2,6%. Καλό μου φαίνεται. Βελτιώθηκαν τα πράγματα. Όμω,. Η διαθωτική πολιτική που είναι το πρόσωπο της Ευρώπης ε, προς τις περιφέρειες ε, έγινε ε, καταστροφή. 5% αντί για 3% πέρυσι. Τι θα πούμε στο φορολογούμενο. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόθεσε αρκετά το αίτημά μας για διαφάνεια. Θέλουμε να μας πείτε, να δημοσιεύσετε σε ποιες χώρες πάνε στραβά τα πράγματα. Εδώ και χρόνια θέλουμε εκθέσεις αναχώρα του συνεδρίου όπου να φαίνεται σαφώς ποιος φταίει. Ναι, ναι. Βεβαίως ε, πρέπει να ε, καταδείξουμε ποιοι φταίνε. Φταίει η γραφειοκρατία βέβαια. Και εμείς φταίμε εάν ε, επιτρέπουμε τελικά να απαιτούνται πληρωμές πολλά χρόνια μετά. Η Επιτροπή και το Συνέδριο αποφεύγουν την ευθύνη. Δεν παρεμβαίνουν. Κρύβονται πίσω από δειγματοληπτικού ελέγχου και στατιστικέ. Όλοι κρυβόμαστε πίσω από την μεικτή διαχείριση και αποφεύγουμε να αναλάβουμε τη δική μα ευθύνη. Θα μπορούσαμε από κοινού να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δώστε μα και στον ίδιο σα την ευθύνη που δεν υπάρχει ακόμη περισσότερη διαφάνεια. Και στα κράτη-μέλη και για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Τα επόμενα χρόνια θα επιμείνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ισνάλφος Γκραπίνη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν κύριε Ελένη για την εξαιρετική σα αυτή έκθεση για το οικονομικό έτος 2018. Λεπτομερέστατη έκθεση και καταδεικνύει πραγματικά την πολυπλοκότητα του ζητήματος εκατοντάδες χιλιάδες ημέρες ελέγχου στις οποίες έχουν αναλωθεί οι συνεργάτες σας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αποδώσει έλεγχοι αυτοί καρπούς. Το βλέπουμε. Συντοποιούμε αυτή τη στιγμή ότι ε, μειώθηκε το ποσοστό διορθώσεων. Το ελεκτικό λοιπόν συνέδριο θα πρέπει να εφαρμόσει μια στρατηγική σύμφωνα με την οποία θα μπορούμε να έχουμε και μια κάποια πρόληψη είναι δικαιολογημένο που και που να εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, θεωρώ, αλλά το καλύτερο είναι να μπορούμε να αποτρέπουμε τα σφάλματα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση βάσει τη πρόληψη. Επίση, 41 ε, μία εκθέσεις έχετε κάνει για του εξωτερικού οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λεπτομερέστατε οι εκθέσεις αυτές και επίση δημοσιεύσατε και πάρα πολλά άλλα συνοδευτικά έγγραφα. Σα συγχαίρω λοιπόν και ω εισηγήτρια για την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα χρησιμοποιήσω και τι δικέ σα εκθέσει. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω κύριε Λένε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι όντως έχουμε μια σημαντική μείωση στο ποσοστό σφάλματος, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Υπάρχουν προβληματικοί τομείο που δεν βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ στους τομείς εκείνους κανονικά θα πρέπει να έχουμε το πιο χαμηλό ποσοστό σφάλματος και είναι πραγματικά θλιβερό ότι για τους τομείς αυτούς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει α, καλή επένδυση των κοινοτικών κονδυλίων. Πολλές φορές εντοπίζουμε μάλιστα και κατασπατάληση. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής για το 2018, εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπήρχαν εταιρείε δικαιούχοι, μάλλον που δεν ήταν δικαιούχοι και που λάβανε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα η νομοθεσία μα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Σίγουρα αυτό από μόνο του μπορεί να οδηγεί σε κάποια σφάλματα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί τελικά να παρακολουθήσει, να ακολουθήσει και να εφαρμόσει τη δική της νομοθεσία εντοπίζουμε περιπτώσεις προβληματικές της προσλήψης σε διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ίδια προβλήματα εντοπίζουμε και όσον αφορά την κατάρτιση του προπολογισμού των θεσμικών αυτών οργάνων. Και εγώ πραγματικά θλίβομαι όταν βλέπω ότι υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα τα οποία κατασπαλα... κατασπαταλώνται με τον πλέον λανθασμένο τρόπο. Χρηματοδοτούμε προγράμματα τα οποία δεν είναι καν επιλέξιμα. Ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτε αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο. Θα πρέπει τα χρήματά του να επενδύονται και να δαπανώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Δύο αιτήματα έχω εδώ και μπορώ να τα δεχθώ και τα δύο. Ο κύριος Πόλτσακ έχει πρώτο το λόγο, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το ελεκτικό Συνέδριο για την έκθεση αυτή που μας δίνει μια πολύ καλή επισκόπηση της κατάστασης και πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την περαιτέρω δική μας εργασία. Ωστόσο, αυτό το οποίο βγήκε από τη συζήτησή μα είναι το ποσοστό σφάλματο. Το ποσοστό σφάλματο ουσιαστικά συνδυάζεται με τι όλε προσπάθειε απλούστευση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διακύμανση από έτο έτο όσον αφορά το ποσοστό σφάλματο. Όσον αφορά τι αγροτικέ επιχειρήσει και τα προγράμματα πρασινίσματο, ξέρετε ότι μια εταιρεία η οποία, γεωργική η οποία θέλει να υποβάλει ένα πρόγραμμα πρασινίσματο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρώσει πάρα πολλά έγγραφα και να μελετήσει ένα ολόκληρο εγχειρίδιο πολυσέλιδο. Και νομίζω ότι δεν δίδονται εδώ πέρα σωστέ πληροφορίε, οι οποίε πολύ συχνά παραπλανούν. Νομίζω ότι θα πρέπει καταρχά να ασχοληθούμε με το ζήτημα των επιδόσεων. Αν τελικά δαπανούμε σωστά τα κοινοτικά κονδύλια και αν έχουμε τι ευκτέ επιδόσει. Ευχαριστώ. Τέλο, ο λόγο πηγαίνει στον συνάδελφο Τσοχοντάρου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μας αρέσει αυτό που έχει πετύχει το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν κάποια πράγματα να βελτιωθούν. Και φυσικά ε, δεν είναι όλα αυτά ε, τέλεια, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη ε, και έτσι ώστε να μπορέσουμε για παράδειγμα να πάμε σε αυτούς που ε, έχουν κάνει τα λάθη και να τους βοηθήσουμε, να δούμε τι πρέπει να γίνει, πώς θα υπάρχει απλούστευση, να φτιάξουμε τα στάνταρα ώστε να μην χρειάζεται πια να διαπράττονται τέτοια σφάλματα. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν... Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος Έτιγκερ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Η απλούστευση, ναι, όντως, ε, συμφωνούμε. Κάνουμε σχεδόν τα πάντα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού όπου ο καθένας να μπορεί να ζητά χρήματα, να τα λαμβάνει και μετά να τεκμηριώνει πώς θα τα πάνε. Σε αυτά ε, ε, είναι ε, πράγματα που συμβαίνουν μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκής ε, διοίκησης ε, και είναι κάτι που πρέπει να αφορά τις επιχειρήσεις, τα σχολεία, τις μη κυβερνητικέ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα απλό εντύπω, να υπάρχει λίγη γραφειοκρατία για να μπορούμε να αποφύγουμε τη διαφθορά και τα λάθη, τα σφάλματα. Όπως και να έχει βέβαια υπάρχουν οι ε, υπερβάσεις. Τα τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο, η πολυπλοκότητα οι περισσότερες διατάξεις, η περισσότερη τεκμηρίωση ήταν μεγάλα θέματα. Με το νέο πλαίσιο μετά το 2020 θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη απλούστευση και αυτό θα πρέπει και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να το έχετε υπόψη σας όταν θέλετε να προτείνετε κάποιες επιπλέον διατάξεις. Η εφαρμογή του προπολογισμού, ο έλεγχος σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο μπορεί να διασφαλίσει την ε, ποιότητα η τακμηρίωση, ε, η αξιολόγηση, η αποφυγή των λαθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι ε, ε, στο ίδιο επίπεδο όπως ε, έχουμε και σε περιφερειακό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Ε, δεν πρέπει η δουλειά μας εδώ να είναι σε χειρότερο επίπεδο από ότι σε, άλλα, σε άλλου, στα κράτη ή στις περιφέρειες. Εντάξει. Ε, λάθη όλοι κάνουμε, αλλά πρέπει να τα διορθώνουμε. Πρέπει να βρούμε και τις ε, βέλτιστες πρακτικές. Ε, πώς ε, θα προλάβουμε τα λάθη, να μάθουμε από τα λάθη των άλλων, να μην επαναλαμβάνονται. βλέπουμε ότι το ποσοστό σφαλμάτων, το 2,6% ε, εμείς ε, θα προσπαθήσουμε ε, να διατηρηθεί, να μείνουμε σε χαμηλά επίπεδα ως Κομισιόν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ένα 2% πολλές φορές μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι αρχίζει μια συγκεκριμένη τάση. Βλέπω μια σειρά από ζητήματα που θύχτηκαν, αλλά δεν βλέπω τους ομιλητές. Είναι η τελευταία μου ευκαιρία να σας το πω. Είναι ε, μια ε, εμπειρία που είχα πάντα να ε, βρίσκομαι εδώ στο κοινοβούλιο, να τίθεται μια ερώτηση σε εμά, επικριτική, σε εμά στο ελεγκτικό συνέδριο και αυτοί που την έκαναν την ερώτηση να φεύγουν να πάνε για καφέ. Όμως αυτό είναι συναδελφικότητα. Ε, είναι μια μορφή ευγένεια σε μια δημοκρατική συζήτηση. Καλό είναι να ακούει κανείς την απάντηση στην ερώτηση που ο ίδιος έχει θέσει. Ε, δεν λέω μόνο για εκείνη την ομάδα των ανθρώπων ε, που έχουν αυτή την πολεμική διάθεση, αλλά και για τον συνάδελφο Λέκα. Το είπε και ο ίδιος, ότι δεν παίρνει απαντήσεις. Κύριε Πίπερ, ε, η πλήρης διαφάνεια το να δίνουμε δεδομένα εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Προσπαθούμε με την διαφάνεια να ε, επιβάλλουμε, να εφαρμόσουμε πλήρως ε, τους κανόνες. Ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Αν θέλει κάποιος παραπάνω, μπορεί κανείς να το ελέγξει. Τα λάθη δεν είναι τόσο διαφανή όσο στην περίπτωση της απάτης ή της διαφάνειας. Εκεί πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένες χώρες και επιχειρήσεις που θα πρέπει να τιμωρηθούν. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, ο κύριος Λένε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς Ευχαριστώ την κυρία Χολμάιερ, πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προβολισμού. Και εμεί χαιρόμεθα για τη συνεργασία μαζί σα, και την Επιτροπή σα κατά τη νέα θητεία. Αναφερθήκατε στο κεντρικό θέμα που το είπαν και πολλοί συνάδελφοι. Όσο πιο περίπλοκοι είναι οι κανόνε, τόσο υψηλότερο το ποσοστό και η πιθανότητα σφαλμάτων. Η βάση λοιπόν του προβλήματος είναι αυτή και προς ε, την πλευρά όλων μας και μου γιατί ήμουν 22 χρόνια ευρωβουλευτής πρέπει να πω ότι είναι η ευθύνη του νομοθέτη. Ο νομοθέτης προκαλεί αυτή την τάση. Όλο και πιο αναλυτικές διατάξεις. Γιατί δεν εμπιστεύεται τη διοίκηση. Προσπαθεί να ρυθμίσει την κάθε μεμονωμένη περίπτωση, όλες τις λεπτομέρειες. Και αυτό ισχύει για όλες τις πλευρές των νομοθετικών σωμάτων, όλα τα όργανα. Κοιτάξτε, τώρα που έχω κάτσει από την άλλη μεριά, βλέπω τι προβλήματα δημιουργούνται στη δίκηση με αυτήν την νομοθεσία. Καλό είναι να εμπιστευόμεθα περισσότερο τη δίκηση και σε ευρωπαϊκό και σε επίπεδο κρατών μελών, ούτως ώστε με σαφέστερους και απλούστερους κανόνες που μπορεί να χρειάζονται ερμηνεία, αλλά παρόλα αυτά θα καταλήξουν σε καλύτερη εφαρμογή. Αυτό είναι το αποφασιστικό. Πρέπει να επιδιώξουμε πραγματικά να βελτιώσουμε αυτή την ε, βασική αδυναμία και θα μειωθούν έτσι και τα σφάλματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όσους επένεσαν τα πιλωτικά προγράμματα και για τον έλεγχο που βασίζεται σε πιστοποιητικά. Τι κάνουμε. Ελέγχουμε και τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και βλέπουμε πόσο θα πάνε καλά, τι ελλείψεις έχουν και μετά σε διάλογο με την Κομισιόν και τις άλλες υπηρεσίες που ελέγξαμε προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να δημιουργήσουμε και κανόνες για το πώς θα τους βοηθήσουμε. Και αυτή η νέα προσέγγιση έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις. Κύριε Σαστέλ, είπατε ότι κάθε χρόνο μιλάμε για τα ίδια προβλήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα ε, η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία. Τα αναφέραμε. Κάτι που είπε η κυρία Γραπίνη και ο κύριος Σαστέλ ε, επικεντρώνουμε όχι μόνο στη συμμόρφωση αλλά και με τη λογιστική ακρίβεια και πρέπει μας είπε να ασχοληθούμε και περισσότερο με την αποδοτικότητα Κοιτάξτε οι εκθέσεις που είχαν να κάνουν με την ε, απόδοση έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια Όντως λοιπόν έχουμε ε, μετακινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι και εσάς και στους πολίτες κυρίως σας ενδιαφέρει εάν η γέφυρα, το αεροδρόμιο, το λιμάνι που οικοδομήθηκαν με ευρωπαϊκούς πόρους ε, χρησιμοποιείται, αν χρησιμοποιείται με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Δεν τους ενδιαφέρει, για παράδειγμα, εάν στην προκήρυξη έγινε ένα τεχνικό λάθος και δόθηκαν ε, λάθος τεχνικά στοιχεία. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι χρησιμοποιείται αυτή η υποδομή. Είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό ίσως και πιο σημαντικό. Η κυρία Φολκραμόν ε, Ταουμπαντέλ και η κυρία Βότερς ε, ασχολήθηκαν με τη βιωσιμότητα. Μα θα είδατε και θα το δείτε όταν θα αποφασίσουμε τη νέα μας στρατηγική για το πώς θα λειτουργήσουμε από το 2021 και μετά. Θα δείτε λοιπόν ότι θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τους ε, στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, με τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους θα είναι ε, βασικό στοιχείο της διαμόρφωσης της δραστηριότητάς μας. Άρα θα σκοτούμε περισσότερο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια ορισμένων συναδέλφων. Σας διαβεβαιώνω ότι, θα το δείτε και τον διαβάσετε την έκθεση, αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα που πήγαν στραβά τα πράγματα. Γιατί η κριτική είναι απόλυτα αναγκαία για να βελτιώσουμε. Το κάνουμε δεκαετίες και θα το συνεχίσουμε. Ο κύριος Τσαριέτσκι, αλλά και ο κύριος Χίβερ και άλλοι είπαν θέματα για τα οποία πρέπει να μιλήσω. Η μέθοδός μας είναι στατιστική. Η συνθήκη μας υποχρεώνει να δώσουμε δήλωση αξιοπιστίας για την εκτέλεση του προπολογισμού συνολικά. Κανείς δεν είναι σε θέση να εξετάσει τα εκατομμύρια πράξεων που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε λεπτομέρεια, κάθε μία. Κάνουμε αυτό που λένε οι διεθνείς ε, προδιαγραφές και που χρησιμοποιούν όλοι οι ε, οργανισμοί ελέγχου παντού. Παίρνουμε πράξεις που να έχουν στατιστικά αξιοπιστία, τις επιλέγουμε κατά τύχη και τις ελέγχουμε. Και με βάση τα αποτελέσματα βλέπουμε ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος. Είναι πολύ απλό σύστημα σε ένα πληθυσμό ας πούμε ε, χιλιάδ, χιλίων για παράδειγμα ε, πράξεων που ελέγξαμε συγκεκριμένα ήταν 750 βρήκαμε ότι 59 είχαν πρόβλημα και μετά έχουμε και ένα περιθώριο σφάλματος αυτοί είναι οι διεθνείς κανόνες με βάση τους οποίους εργαζόμεθα και μπορούμε βεβαίως να κάνουμε πιο ακριβείς να γίνουμε πιο ακριβείς μπορούμε να ασχοληθούμε με πολύ περισσότερε λεπτομέρειε. Υπάρχουν πολλέ δευτερεύουσε πλευρέ του προπολογισμού. Αλλά να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερου πόρου. Πολύ περισσότερου. Αυτή τη στιγμή οι μισοί πόροι μα πηγαίνουν σε αυτού του ελέγχου. Στα πλαίσια τη ετήσια έκθεση. Αν θέλουμε να γίνουμε ακριβέστεροι, αυτό σημαίνει, κοιτάξτε, αυτά είναι μαθηματικά. Για να έχουμε διπλή ακρίβεια, θέλουμε τετραπλού πόρου. Έτσι είναι. Το, συμβούλιο, ε, το, το συνέδριο συγγνώμη, έχει τώρα γύρω στου ε, χίλιου υπαλλήλου. Αν μα δώσετε 4.000 υπαλλήλου, θα έχουμε διπλό ποσοστό ακρίβεια. και διπλές πληροφορίες. Αυτό είναι το αποφασιστικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με αυτούς που αποφασίζουν τον προπολογισμό. Με τους πόρους που έχουμε περιοριζόμαστε σε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Και για να αξιοποιήσουμε σωστά τους πόρους, κάνουμε μια εκτίμηση κινδύνου. Ελέγχουμε περισσότερο εκεί που ξέρουμε ότι υπάρχει και μεγαλύτερος κίνδυνος. Εκεί που έχουμε διαπιστώσει μέσα από δεκαετίες ελέγχου, ελέγχου ότι είναι χαμηλό το ποσοστό σφαλμάτων σε κάποιες διοικήσεις, εκεί φυσικά κάνουμε λιγότερους ελέγχους. Προσπαθούμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε σωστά τους πόρους μας, ούτως ώστε να έχετε κι εσείς το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι απάντησα στην ερώτηση της κυρίας Γκαρσία για τις στατιστικές μεθόδους. Ο κύριος Μπόγιε είπε η ποσότητα των πόρων μας. Κοιτάξτε, στις ε, προτάσεις για το πολιετές πλαίσιο έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και εμείς. Μπορείτε να τις διαβάσετε. Ο κύριος Νόβακοφ ασχολήθηκε με την ε, αποδοτικότητα. Είπαμε ότι έχουμε αλλάξει το κέντρο βάσμα. Ο κύριος Γιούτσικα αναφέρθηκε στις δημοσιεύσεις του ΩΣΑ. Όντως πιστεύουμε ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ υψηλό επίπεδο εκτέλεσης του υπερπολογισμού. Πολύ καλές προδιαγραφές, πολύ καλό επίπεδο έχουμε βέβαια. Πάντα μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Το είπαμε, αναμφίβολο. Τα γράφουμε και στην έκθεσή μας. Αλλά αν ε, συγκρίνουμε παγκοσμίω Υπάρχει για παράδειγμα το Γραφείο των Πολιτείων. το Γραφείο για τη Λογοδοσία των Κυβερνήσεων, που κάνει κάποιε συγκρίσει. Και εκεί είμαστε σε πολύ καλή θέση. Το Government Accountability Office. Να σκεφτούμε πού ήμασταν. Το 1990 η Επιτροπή του Ζαν Κατσαντέρ παρετήθηκε. Χρειάστηκε να παρετηθεί. Και τότε έκανε και τότε εκθέσει στο Ελεκτικό συνέδριο. Οι ε, εκθέσει αυτέ ε, έδιναν αρνητική πιστοποίηση στον προπολογισμό. Τότε, στη δεκαετία του 90, δεν δημοσιεύαμε στοιχεία για διάφορα τμήματα του προπολογισμού. Γιατί είχαμε σφάλματα διψήφια. Η κατάσταση τότε ήταν ότι δεν υπήρχαν ε, λειτουργικά εσωτερικά συστήματα ελέγχου των θεσμών. Αν τα συγκρίνουμε όλα αυτά με τη σημερινή κατάσταση, τότε έχουν σημειωθεί τρομερές πρόοδοι. Και πρέπει να το πω. Και χάρη και σε εσά έγινε αυτό. Διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το 1999 έκανε σημαντικέ αλλαγέ στον δημοσιονομικό κανονισμό και υπήρχε πάντα επίση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού και επίση μα έδωσαν του πόρου για να μπορέσουμε να κάνουμε τι αλλαγές που κάναμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν ουσιώδει πρόοδοι. Κάτι για τον κύριο Πίπερ. Είναι το ίδιο που είπα και προηγουμένω. Με άλλο τρόπο. Φυσικά, θεωρητικά, θα μπορούσαμε να σα δώσουμε στοιχεία για τι χώρε, αλλά τότε θέλουμε περισσότερου πόρου όταν ελέγχω 750 ή 800 πράξεις συνολικά για τον προπολογισμό. Για ορισμένε χώρε τι έχω. 16 πράξεις για παράδειγμα ελέγχω για κάποια χώρα. Στατιστικά είναι απόλυτα αμεληταίο. Δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, είναι σαν μια δημοσκόπηση. Αν ρωτήσετε χίλια άτομα, έχετε ένα λογικό αποτέλεσμα όσον αφορά, για παράδειγμα, το αποτέλεσμα των εκλογών. Αν ρωτήσετε μόνο 16 άτομα, τότε τι, αποτέλεσμα θα βγάλετε για τι εκλογέ. Αυτό κάνουμε κι εμεί. Σε αντίδραση ε, στις επιθυμίες του Κοινοβουλίου τι κάναμε. Κάθε 7 χρόνια, το κάναμε για πρώτη χρονιά το 2014, πρώτη φορά το 2014, όλα τα στοιχεία που είχαμε για τα προηγούμενα χρόνια τα δημοσιεύσαμε. Αλλά με μια καθαρή προειδοποίηση ότι τα στοιχεία, αυτά δεν έχουν στατιστική σημασία. Δεν έχουν στατιστική αξία για την αξιολόγηση της κατάστασης σε κάποιο κράτος μέλος. Σε αυτό το σημείο είμαστε και δεν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θα σας πω αυτό που είπα και στο ΕΚΟΦΗΝ πριν από δύο εβδομάδε. Γιατί και από το Συμβούλιο έχω διάφορε επιθυμίε ε, περισσότερα εδώ, περισσότερε λεπτομέρειε εκεί, για τον τάδε κλάδο. Με του πόρου που έχουμε δεν το μπορούμε. Και όσε φορέ και να μα το ζητήσετε δεν είναι εφικτό. Εκτό αν ε, μα δώσετε και άλλου πόρου. Αλλά παρόλα αυτά θα είχε έννοια οικονομικά να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε τόσο περισσότερου πόρου για, για να χρησιμοποιήσουμε σε τόσο διαφορετικού τομεί του προπολογισμού. Αλλά είναι δική σα απόφαση. Δική σα η απάντηση. Όχι εμεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η συζήτηση κλείνει. Ολοκληρώνεται. Επόμενο θέμα προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για να συμμετάσχετε στο Catch the ή για να γύρετε μια μπλε κάρτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ε, την κάρτα ψηφοφορίας που έχετε, τη χρειάζεστε δηλαδή. Για το ΚΑΤΣΙΑΙΤΑ θα το κάνετε τώρα χωρίς να περιμένετε μέχρι το τέλος της συζήτησης. Και τώρα ο πρώτος που θα μιλήσει είναι ο εισηγητής της ερώτησης. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που σας ε, παρουσιάζω ε, το, ένα ερώτημα για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Την έρευνα και την διάσωση στην Μεσόγειο. Την έρευνα και διάσωση ανθρωπίνων ζωών έναντι ε, του αφόρητου φόρου που, θανάτου που πληρώνουμε τόσα χρόνια για αυτό το θέμα. Το έχουμε πει τόσες φορές εδώ στο Στρασβουργό. Θα κάνω κάποιες παρουσια... παρατηρήσεις στα αγγλικά σύμφωνα με το έγγραφο που έχει κυκλοφορήσει μετά από τη συζήτηση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και μετά θα περάσω στα ισπανικά για να μπορέσω να κάνω κάποιες τελικές ε, δηλώσεις. Ε, το να παρουσιάζει κανείς ε, το θέμα αυτό στην ουσία δείχνει και τη σημασία του ιστορικού αρχείου ας πούμε που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε φορά που υπάρχει μια τραγωδία στη θάλασσα, στη Μεσόγειο, χίλιες ζωές για παράδειγμα χάνονται, σχεδόν τελετουργικά κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μας λυπεί η τραγωδία αυτή. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τα δεδομένα. Καλούμε Επιτροπή και Συμβούλιο για ανάληψη πραγματικής δράσης επί του θέματος. Αυτός είναι ο σκοπός του ψηφίσματος. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε όλα τα σημαντικά θέματα που έθεταν οι ομάδες του Κοινοβουλίου για να περάσει το μήνυμα, να φτάσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και να δείξουμε ότι μας νοιάζει η ανάγκη αυτή να σταματήσουν οι θάνατοι στη θάλασσα. Πολλές ζωές χάθηκαν γιατί δεν υπάρχει τρόπος να φτάσουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό εκτίθενται στην εμπορία, ε, του στην εμπορία τους και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους παραβιάζονται. Παραβιάζονται και στις πατρίδες τους, στη Λιβύη Άρα λοιπόν δεν λέμε ότι υπάρχει μόνο ανάγκη να βελτιωθούν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, τα νόμιμα μέσα, αλλά να, καλέσω, να, να ονομάσουμε την Λιβύη με το όνομά της. Δεν είναι ασφαλής. Μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε τις την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα με την Frontex, σε συνεργασία με κάποια κράτη-μέλη και σε συνεργασία με την ακτοφυλακή της Λιβύης. Οι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν όμως υπόκεινται στις λιβιακές αρχές που, θεωρούν, που τους θεωρεί ε, εγκληματίες διότι παρατύπως εγκαταλείπουν το έδαφος. Και δεν τους δίνει την ευκαιρία να φύγουν νομίμως. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που επιστρέφουν στη Λιβύη θα ε, υπαχθούν σε μεγάλη καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Και δεν θέλουμε να είμαστε συνεργοί σε κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, μια, ένα νομικό επιχείρημα, το οποίο ακούστηκε στις ε, συζητήσεις. Η ανάγκη να αποποινικοποιηθούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που σώζουν ζωές εκεί, που συνεργάζονται για να σωθούν ζωές. Βεβαίως, σεβόμεθα τις προσπάθειες που έγιναν από τις δημόσιες αρχές στην Ιταλία, την Ισπανία, όπου επένδυσαν πολλά δημόσια κονδύλια για να ε, αντιμετωπίσουν το θέμα ως οι νότιες ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως, σώζονται ζωές, αλλά ε, και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα πρέπει να κινηθούν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο με τρόπο που θα συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο. Και όταν μιλώ για ενωσιακό δίκαιο, μιλώ και για διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο το οποίο διακυβεύεται, διότι οι αρχές αυτές ε, είναι και δικές μας σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, που τέθησαν σε ισχύ πριν από 9 χρόνια. Ε, υπάρχει παραβίαση του άρθρου 18, για παράδειγμα, το δικαίωμα να ζητήσει κανείς άσυλο. Τώρα χρειάζεται ε, να έχουμε μια απάντηση προς τους ετούντες άσυλο ως Ευρωπαίοι με τρόπο που θα συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες, αρχές και σημαίνει βεβαίως υπευθυνότητα, και επιμερισμένη ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά υπάρχουν. Εμείς καλούμε την Επιτροπή με το Συμβούλιο να κάνει μια νέα αρχή, με νέα εντολή, να ξεμπλοκάρει το, τη δέσμη του ασύλου θα πρέπει να ε, επανεξεταστούν ε, κάποιες επίμαχες διατάξεις, να σταματήσει η ποινικοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, να ανοίξουν τα λιμάνια στα σκάφη που έχουν σώσει στην ανοιχτή θάλασσα ζωές σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Γιατί η ε, σύμβαση του δικαίου της θάλασσας της Ιαμαϊκής το 1982 και οι συμβάσει για την διάσωση στη έρευνα και διάσωση ε, ε, εξακολουθούν να δεσμεύουν όλα τα κράτη-μέλη, όπως δεσμεύουν και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο απάντησης, λοιπόν, που να έχει νόημα. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ψηφορία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο την Πέμπτη, να καταδείξει την ίδια βούληση να ενισχύσει το μήνυμά του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή που έδειξε σε προηγούμενα ψηφίσματα. Συγκεκριμένα το ψήφισμα που ενέκρινε ε, τη λεγόμενη ολιστική προσέγγιση, μια περιεκτική θεώρηση του προσφυγικού και του συστήματος χορήγησης ασύλου. Ε, αυτή τη στιγμή κυρία Μετσόλα από το ΕΛΚΑ και η κυρία Σεσίλια Κέγκε από τους Σοσιαλιστές ε, εργάστηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο παραμένει κρεμές το, εντολή την οποία ανέλαβε το Κοινοβούλιο να τερματίσει την ποινικοποίηση των ΜΚΟ που εργάζονται σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει λοιπόν το μήνυμα αυτό να ανανεωθεί με ιδιαίτερη έμφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η κυρία Τούπουράινεν έχει το λόγο. Ξεκινώντας, θα πω ότι η κατάσταση στη Μεσόγειο εξακολουθεί να μας ανησυχεί. Βέβαια θα παρατηρήσει κανείς ότι έχουν υπάρξει σοβαρές βελτιώσεις 170.000 πέρασαν από τους τρεις δρόμους της Μεσογείου το 18. Είμαστε 20% χαμηλότερα για την αντίστοιχη περίοδο φέτος. Αλλά παρόλα αυτά έστω και ένας θάνατος δυστυχώς είναι απαράδεκτος. Έχει μειωθεί βέβαια κατά 44% σε σχέση με το 18 το οποίο αποδίδεται και στη μείωση των αναχωρήσεων και στην αύξηση των ικανοτήτων της Λιβικής Ακτοφυλακής. Από τις αρχές Οκτωβρίου 688 έχασαν τη ζωή τους, πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν την Νότια Μεσόγειο. Είναι μια τραγωδία, ακόμα και αν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζουν ότι το 18 η, Λιβική ακτοφυλακή ε, παρά την δύσκολη κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη έσωσαν πολύ κόσμο και ήδη έχουν σώσει μέχρι τώρα 7.800. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν τη σημαντική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει τις τραγωδίες αυτές. Ιδιαίτερα προς τη Λιβύη η βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω της έλλειψης πόρων του Λιβυκού κράτους. 91,3 εκατομμύρια προς τη Λιβυκή ακτοφυλακή και επίσης την δημιουργία συντονιστικού κέντρου διάσωσης στην χώρα αυτή. Ε, η επιχείρηση Σοφία έχει δώσει την δυνατότητα για την εκπαίδευση 3.000 στελεχών όπως επίσης και ε, παρά τις τρεις τελευταίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο που έσωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές η βοήθεια η οποία δίδεται είναι σημαντική στις χώρες της Βορείου Αφρικής, αλλά η κατάσταση στον τομέα της έρευνας και διάσωσης δεν είναι ικανοποιητική. Υπάρχει έλλειψη ευθυνών, υπάρχει έλλειψη κατανομής των υποχρεώσεων και των ευθυνών, δεν υπάρχει σωστός σεβασμός του θαλασσίου δικαίου απαιτείται πιο στενή συνεργασία ε, στο SAR με τους εταίρους μας. Αυτό δεν είναι μόνο μία ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο ε, είναι υποχρεωτικό για όλες τις χώρες. Για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε λοιπόν τους εταίρους, τους εταίρους μας να φέρουν εις πέρας την υποχρεώ, τις υποχρεώσεις τους, βοηθάμε χώρες όπως το Μαρόκο, την Ισία, Αίγυπτος ε, και στα πλαίσια της ε, διαχείρισης των κινδύνων και στα πλαίσια της στήρησης και του σεβασμού του διεθνούς ε, δικαίου της θάλασσας. Ξέρετε ότι έγινε μια αλλαγή που επιτρέπει πλέον να να έρχονται σε, στα λιμάνια τα Ιταλικά, τα πλοία διάσωση στον Μικείο από ε, την ε, Νότια Μεσόγειο ε, για να υπάρξει σωστή διαχείριση αυτών των αφήξεων από το καλοκαίρι τα κράτη-μέλη προσπαθούν να βρουν μια κοινή λύση. Στις 31 Σεπτεμβρίου έγινε μια κοινή δήλωση για ένα μηχανισμό ο οποίος θέλει να αντικαταστήσει τον κανονισμό που ισχύει σήμερα μεταξύ ε, Βελγίου, Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας. Εν μεταξύ και κάποιες άλλες χώρες συμμετέχουν και κάποιες άλλες προσκλήθηκαν να συμμετέχουν. Είμαι πεπισμένη ότι αν ο μηχανισμός αυτός εργαστεί σωστά, τότε πραγματικά θα είναι το καλύτερο κίνητρο για να συμμετέχουν όλες οι χώρες οι χώρες οι οποίες στο παρελθόν ε, εδέχονται ε, μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών από τη Μάλτα και την Ιταλία ε, συζητούν σήμερα κάποιες διαδικασίες πιο δεσμευτικές. Ακόμα όμως και αν ο μηχανισμός αυτός είναι αποτελεσματικός, δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός μας στόχος. Πρέπει να βρούμε μία μακροπρόθεσμη λύση στην κατάσταση αυτή, και γενικότερα στο σύνολο των προβλημάτων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χορήγησης Ασύλου. Απαιτείται να υπάρξει μια αηφόρος λύση που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην σωστή κατανομή των ευθυνών. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί και σε περιπτώσεις κανονικής θα έλεγα εξέλιξης του φαινομένου και σε περιπτώσεις κρίσεων να είμαστε καλύτεροι στον έλεγχο αυτών ε, οι οποίοι έρχονται στην Ένωση και να επιστρέφουμε στις χώρες τους αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα και που δεν έχουν, δεν, ε, αν θα έλεγα εκπληρούν τις προϋποθέσεις ε, για τη χορήγηση ασύλου. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν όμως με συνολικό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επιτρέψει νομίζω την αποκατάσταση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και να αποτελέσει και τμήμα του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι πρόκειται για τη συνέχεια των προτάσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν και καλείται η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα εξετάσει. Στα πλαίσια τώρα της ποινική δίωξης των οργανώσεων που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, ο ρόλος των μικιών δεν μπορεί να αγνοηθεί, όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Λίμπε. Και όπως μας υπενθυμίζει με το ψήφισμά του το Κοινοβούλιο, το ψήφισμα του μηνός Ιουλίου του 19, οι οργανώσεις αυτές σώζουν ζωές στην ανοιχτή θάλασσα. Απαιτείται λοιπόν οι κυρώσεις να υπάρχουν όταν υπάρχουν κίνδυνοι, ε, θα έλεγα, ποινικής, ποινικά κολάσιμης δράσης από αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή μόνο. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, προς τα κράτη-μέλη έτσι ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια, η γνήσια να μην διώκεται με οποιοδήποτε τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Χάν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Ε, τα τελευταία χρόνια εφαρμόσαμε μια περιεκτική πολιτική μετανάστευσης και χάρη σε αυτήν ε, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις τις οποίες θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε ε, συνολικά με θετικό τρόπο. Η κατάσταση της ε, μετανάστευσης έχει μειωθεί και έχει επανέλθει σε προηγούμενα επίπεδα. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή ε, ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει ο, ενώ ο αριθμός των ε, νεκρών στη Μεσόγειο έχει μειωθεί, παρόλα αυτά παραμένει υψηλός. Η κάθε μεμονωμένη απώλεια ε, συνιστά μια τραγωδία, ενώ από τις θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Χαίρομαι που έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να συζητήσουμε το σημαντικό θέμα της έρευνας και της διάσωσης ανθρώπινων ζώων στη Μεσόγειο. Η διάσωση ήταν πάντοτε προτεραιότητα της ε, Κομισιόν. Από το 2015 730.000 άνθρωποι διασώθηκαν στη θάλασσα. Οι τρεις από αυτές τις επιχειρήσεις συντονίστηκαν από την ακτοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την επιχείρηση Σοφία, οι χώρες μέλη ε, συμφώνησαν να συνεχίσει ε, ε, η δέσμευσή μας ε, να διασταθούν ε, ζωές δεν ξεκινάει μόνο όταν οι άνθρωποι αυτοί φτάσουν στα σύνορά μας. Η πρόληψη επίσης περιλαμβάνει μέτρα για να υποστηριχθούν οι πρόσφυγες στις τρίτες χώρες πριν ξεκινήσουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι. Όταν μιλάμε για έρευνα και διάσταση θα πρέπει να λησμονούμε ότι εμπίπτει ε, αυτή στην αρμοδιότητα των χωρών μελών στη βάση του διεθνού δικαίου της θάλασσας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την δυνατότητα να συντονίζει αυτές τις δραστηριότητες και για τον ίδιο λόγο δεν έχουμε το δικαίωμα ή το καθήκον να παρεμβαίνουμε. Ε, αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Ε, αλλά ε, έχουν το καθήκον βεβαίως να συνδράμουν ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Αυτό με φέρνει στο ζήτημα της ε, διευκόλυνσης που παρέχουν ορισμένοι άνθρωποι, τους οποίους δεν θα έπρεπε να ποινικοποιούνται. Καμία μορφή συνδρομής προς τους πρόσφυγες που βρίσκονται σε απόγνωση, αντιμετωπίζουν δυσχέρειε στις, ε, στα νέα εδάφη που βρίσκονται θα πρέπει να ποινικοποιούνται. Και αυτοί ωστόσο αυτοί οι οποίοι διασώζουν τα άτομα αυτά θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές ε, δίκαιο. Ε, μία εγκεκριμένη είσοδος ε, σε μία χώρα βεβαίως δεν δίνει καμία λαβή στην ποινικοποίηση των, της δραστηριότητας συνδρομής προς τους ανθρώπους αυτούς. Η αξιολόγηση της Επιτροπής του Νομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2017 αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σαφήνεια στην εφαρμογή των νόμων ανθρωπιστικής, εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους. Σαν αποτέλεσμα, εξολόγηση αναγνωρίζει την ανάγκη οι χώρες μέλη να έχουν ένα διάλογο με τις ΜΚΟ προκειμένου να διευκολύνουν τη συνεργασία, να διευκρινίζουν τα περιεχόμενα και να ασχολούνται με τις ανησυχίες που συνδέονται με την ποινικοποίηση. Επίσης, η Επιτροπή ε, έρχεται σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να έχει περισσότερα στοιχεία και να ενισχύσει η διαδικασία εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Η τελευταία συνάντηση έλαβε χώρα την 1η Οκτωβρίου. Τα αποτελέσματα του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών θα δημοσιοποιηθούν. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η Επιτροπή εργάζεται άκουνα προκειμένου να εξεύρει μια λύση όσον αφορά την κατανομή των ανθρώπων που έχουν διασωθεί στη θάλασσα σε συμφωνία με την βασική αρχή της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού της ευθύνης μεταξύ των χωρών μελών. Κατόπιν αιτήματος των χωρών μελών, η Κομισιόν διδραμάτισε ένα καθοριστικό ρόλο ε, σε 15 περιστάσεις ε, πάνω από χίλια άτομα ε, τα οποία αποβιβάστηκαν αυτές τις επιχειρήσεις ε, μετέβησαν ασφαλώς σε άλλες χώρες όπως είναι η Νορβηγία. Ε, βεβαίως η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων αυτών ακόμα δεν έχει μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα. Χώρες όπως η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβανία, η Ισπανία η Γερμανία και λοιπά και άλλες χώρες έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά οφείλονται στο συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής σε συνεργασία με τις χώρες μέλη ε, στη βάση της επιθυμίας της να επιδείξει ελεγγύη όσον αφορά την ε, διαδικασία εγκατάστασης των ε, προσφύγων. Η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει με έμφαση τις χώρες ε, μέλη σε προσωρινά, για προσωρινά μέτρα όσον αφορά την ε, διαδικασία αποβίβασης αυτών των ατόμων ε, και εκπονήθηκε ένας προσωρινός μηχανισμός αλληλεγγύης στον οποίο συμμετάσχει και η Γερμανία και η Μάλτα στην Επιτροπή Δικαιοσύνης και Εξωτερικών Υποθέσεων θα συνεχίσει ο διάλογος με, για τα θέματα αυτά. Ε, οι χώρες μέλη που συμμετέχουν στην υποδοχή των προσφύγων ε, θα ε, συνεχίσουν τις επαφές τους και με την Νορβηγία. Ε, αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι διευθυντήσεις δεν μπορούν παρά να είναι ένα μεταβατικό στάδιο ε, προς την, έως το σύστημα χορήγησης ασύλου. Ε, αυτά βέβαια σχετίζονται με την οδηγία περί επαναπατρισμού και την σχετική με την προστασία των εξωτερικών συνόρων μας ε, σε συνεργασία με τρίτες ε, χώρες που βρίσκονται στις ε, μεταναστευτικές οδούς. Ευχαριστώ πολύ. Για να αρχίσουμε τη συζήτηση και πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, παρακαλώ να τηρείτε τα χρονικά περιθώρια. Πρώτος ομιλητής, πρώτη ομιλήτρια ή εκπρόσωπος της ομάδας ΕΛ και η κυρία Ντυπον. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι υποχρέωσή μας η διάσωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Γι' αυτό συμμετείχαμε στις ε, συζητήσεις για το ψήφισμα. Δεν θέλουμε όμως να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα βοηθάει τους διακίνητες. Δεν θέλουμε να υποστηρίζεται αντί να καταπολεμείται αυτό το κοινικό μοντέλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η, τα αίτια της φυγής βρίσκονται στη στεριά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια διαδικασία διάσωσης, έρευνας και διάσωσης που θα τηρείται από όλους. Χρειάζονται εντατικές συζητήσεις με τις χώρες ε, διέλευσης, τις χώρες προέλευσης ε, και πρέπει να συνεννοηθούμε για τον κοινό αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειάζεται διαφοροποίηση μεταξύ οικονομικών μεταναστών και προσφύγων και για το άσυλο Χρειαζόμαστε ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ε, οι χώρες αυτές πρέπει να υποστηριχθούν. Αυτό που θέλουμε δεν αναφέρεται στο ψήφισμα. Όλα αυτά χρειάζονται όμως για να πετύχουμε τον ύψιστο στόχο να αποτρέψουμε τους ανθρώπους να αρχίσουν αυτό το δρόμο, τον επικίνδυνο δρόμο της φυγής. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σώσουμε ε, περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστώ πολύ. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει ο κύριος Μωράεσε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συνεχιζόμενη κατάσταση στη Μεσόγειο μας θυμίζει τις ευρωπαϊκές αξίες οι οποίες προσβάλλονται πλέον σε καθημερινή βάση. Πρέπει να δράσουμε και νομίζω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Λίμπε είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή να συνδυάσει τις απόψεις των ε, μελών του Κοινοβουλίου γύρω από το θέμα. Νομίζω ότι η ομιλία του δείχνει το τι ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη ή θα κάνουμε κάτι τώρα ή θα αποτύχουμε πλήρως. Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα φαινόμενα αυτά. Πρέπει να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει να ανταποκριθούμε λόγω των αξιών οι οποίες μας χαρακτηρίζουν και ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί οι οποίοι ασκού, ασκούν την έρευνα και διάσωση φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διώκονται ποινικά. Ξέρω ότι το πακέτο μέχρι τώρα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή έχουν, έχει παγώσει, θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε γρήγορα, να υπάρξει λειτουργική συνεργασία, να υπάρξει διαφάνεια για τις δραστηριότητες του Frontex στη θάλασσα και ε, στην στήριξη επίσης των ακτοφυλακών χωρών όπως το Μαρόκο, η Τουρκία, η Αίγυπτος, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σημεία ελέγχου και τέλος τα κράτη-μέλη τα ίδια θα πρέπει να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τις ηθικές τις οποίες έχουν και σε σχέση με την έρευνα και διάσωση ε, συνεργαζόμενοι και με τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στις περιοχές τους. Το ψήφισμα αυτό από τη μία δείχνει το τι μπορεί να κάνει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη τα κράτη-μέλη γιατί για τα κράτη-μέλη αυτό το blame game, αυτή η κατηγορία, η ανταλλαγή κατηγοριών από το ένα στο άλλο κράτος δεν μας οδηγεί πουθενά. Πρέπει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις, αποφάσεις όμως οι οποίες θα είναι οι σωστές αποφάσεις ηθικά και δεοντολογικά και στη Μεσόγειο και γενικότερα. Πρέπει να υποστηριχθεί το ψήφισμα αυτό Ζητάμε τη μέγιστη δυνατή στήριξη έτσι ώστε να μοιραστούμε όλοι τις ανθρώπινες ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ. Από το Ρηνιού η κυρία Ιντβέλτ έχει το λόγο. Πρόεδρε, Υπουργέ, Επίτροπε, ξεκινώντας να πω ότι κάθε ζωή έχει τη δική της αξία. Και όταν μιλάμε για αριθμούς αυτών που πνίγονται στη Μεσόγειο, μιλάμε για ποιους, μιλάμε για ανθρώπους. Ανθρώπους που γεννήθηκαν κάποια στιγμή στον κόσμο αυτό και για τους οποίους οι γονείς τους είχαν ελπίδες. Είναι άνθρωποι σαν και εσάς, σαν και εμένα που ε, δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, το ψήφισμα αυτό έχει να κάνει με την έρευνα και την ανάπτυξη. Δεν έχει να κάνει με ένα ευρύτερο πακέτο για το άσυλο κτλ. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε ώσπου να ολοκληρωθεί το πακέτο για το άσυλο γιατί ο κόσμος εξακολουθεί να πνίγεται. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διάσωσης στη Μεσόγειο. Και αν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτό που πρέπει, τότε είτε εμπορικά πλοία είτε η ΜΚΟ αναλαμβάνουν δράση και δεν θα πρέπει να διώκουμε ποινικά αυτοί, αυτούς οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να σώζουν ζωές λέτε να ξεχωρίζουμε τους οικονομικούς μετανάστες από ε, τους πρόσφυγες δεν έχει σημασία στην παρούσα φάση αυτό πρέπει πρώτα να τους σώζουμε για να καταλάβουμε τι είναι ο καθένας Λοιπόν, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις ε, και νομίζω ότι η Συμφωνία της Μάλτα είναι ένα πρώτο βήμα έτσι ώστε όλα τα κρατημέλη να προσυπογράψουν την προσπάθεια αυτή και από τις 28 χώρες μόνο 4 το έχουν κάνει. Αυτό είναι μεγάλη ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, είναι, ε, λένε ότι δεν είναι κάτι που έχει σχέση με την διάσωση των ε, προσφύγων αλλά όταν πρόκειται για τη διάσωση των προσφύγων τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι παρόντα. Αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκές αξίες, αναφερόμαστε σε χριστιανικές αξίες και σε κάποιες από τις τροπολογίες. Όταν μιλάμε ε, Ε, ο ίδιος για χώρες όπως η Λιβύη και τα λοιπά, ο ίδιος ο πρέσβης της Γερμανίας στη Λιβύη έστειλε μια επιστολή στην Καγκελάριο λέγοντας ότι σε σχέση με τη μετανάστευση η Λιβύη είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και μόνο. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Πρασίνων τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μάκατ. Ευχαριστώ. δεν θα πρέπει να θυσιάζουμε ανθρώπους ε, στον ανθρωπισμό. Και αυτό κάνουμε, αν δεν δώσουμε ένα τέλος στους μαζικούς θανάτους στη Μεσόγειο. Θα πρέπει και με το ψήφισμα να δείξουμε στην Κομισιό να κάνει κάτι παραπάνω και να μην λέει απλώς ότι κανείς δεν πρέπει να χάνει τη ζωή του ε, κατά τη φυγή. Ε, Βέβαια οι τρόποι που επιλέγουν είναι επικίνδυνοι. Δυστυχώς βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η πρακτική. Άνθρωποι που κάποτε ήταν πολύ σημαντικοί για, για, για άλλους. Δεν ε, αποστέλλονται σκάφη ε, διάσωσης. Ε, οι, τα δικαστήρια απαγορεύουν την επιστροφή και τώρα ε, πληρώνουμε την Λιβιακή πολιτοφυλακή να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Ντροπή μας ως Ευρωπαίοι. Πρέπει να υπάρξει μια αποστολή, θα πρέπει να σταματήσει η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, τα αεροπλάνα της Frontex θα πρέπει να ενημερώνουν όλα τα γειτονικά πλοία για να σώζουν τους ανθρώπους αυτούς.